για το οικονομικό έτος 2012. Ε, θα ψηφίσουμε με ονομαστική ψηφοφορία. Θα ήθελε το λόγο η συγγήτρια. Wysoka Izbo, pozwalam sobie zabrać głos, ponieważ nie mieliśmy debaty na temat e, tego budżetu korygującego. Ζήτησα το λόγο γιατί δεν έγινε ουσιαστική συζήτηση και αυτό το θέμα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Η χρηματοδότηση δηλαδή των κοινωνικών δράσεων υπέρ των μεταναστών. Θα ήθελα, συνάδελφοι, να υποστηρίξετε την έκθεση αυτή, γιατί είναι πολύ σημαντικό θέμα για τη μελλοντική χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ πολύ. Ψηφίζουμε με ονομαστική κλίση, η οποία και αρχίζει. Το Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Σας ευχαριστώ πολύ. Κυρία Γέντρε Γεύσκα, εγκρίθηκε με μεγάλη πλειοψηφία η έκθεση. Τώρα έχουμε την δεύτερη έκθεση, την έκθεση Ματέρα, για την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην παγκοσμιοποίηση, με ονομαστική η οποία και αρχίζει, με ονομαστική κλίση. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας της ψηφοφορίας. και πάλι εγκρίθηκε με μεγάλη πλειοψηφία. Το επόμενο θέμα, η επόμενη έκθεση και πάλι της κυρίας Ματέρα αφορά το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση και την αίτηση της, των Ansberg και Düsseldorf αυτοκινητοβιομηχανία στη Γερμανία. Αρχίζει η ψηφοφορία με ονομαστική. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας και πάλι εγκρίθηκε με μεγάλη πλειοψηφία. Τρίτη έκθεση της κυρίας Ματέρα για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση. Ονομαστική ψηφοφορία και πάλι. Ψηφίσατε όλοι. πέρα της ψηφοφορίας. Εγκρίθηκε. Σας ευχαριστώ πολύ. Να ευχαριστήσουμε την κυρία Ματέρα για τις τρεις εκθέσεις της. Στη συνέχεια έχουμε την ε, έκθεση Μορέιρα σε σχέση με την ανταλλαγή επιστολών Ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχές εγκρίθηκε η σύσταση Μορέιρα. Επίσης, έκθεση Μορέιρα, συμφωνία υπομορφή ανταλλαγής επιστολών υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Και η τρίτη έκθεση και πάλι του κυρίου Μορέιρα σε σχέση με συμφωνία μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Νέας Ζηλανδίας υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε τον κύριο Μορέιρα για τις τρεις εκθέσεις. Κυρίες και κύριοι, τώρα περνάμε στην έκθεση της κυρίας Βόρτμαν Κόλ σε σχέση με την εποπτεία της δημοσιονομικής κατάστασης και εποπτεία και συντονισμό οικονομικών πολιτικών. Περνάμε στον κανονισμό. Τροπολογία 13 με ονομαστική κλίση η οποία και αρχίζει. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίθηκε η τροπολογία. Τώρα περνάμε την τροποποιημένη πρόταση με ονομαστική ψηφοφορία. Αρχίζει η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Και πάλι εγκρίνεται. Τώρα ψηφίζουμε το σχέδιο νομοθετικής πρότασης με ονομαστική κλίση η οποία και αρχίζει. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίθηκε. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε και τα συγχαρητήριά μας. Ευχαριστώ, θα ήθελα να συγχαρώ την εισηγήτρια, την κυρία Βόρτμαν Κόλ. Περνάμε στην επόμενη έκθεση, έκθεση της κυρίας Σιλβί Γκουλάρ για τη δημοσιονομική εποπτεία στη ζώνη του ευρώ. Η επόμενη έκθεση, όπως σας είπα, είναι η έκθεση της κυρίας Γκουλάρ για την ε, δημοσιονομική εποπτεία στη ζώνη του ευρώ. Και η Επιτροπή θα ήθελε να λάβει το λόγο για την ε, εποπτεία στη ζώνη του ευρώ. Έχετε το λόγο. Thank you. Ευχαριστώ Πρόεδρε, αγαπητά μέλη. Μπορώ να σας επιβεβαιώσω ότι η δήλωση της Επιτροπής ε, αντικατοπτρίζεται στην τροπολογία 11, αλλά επειδή πρόκειται για μια πολύ σημαντική δήλωση θα ήθελα να σας τη διαβάσω. Πριν από το τέλος του 2011 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα υποβάλει μία έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο για την σύσταση ενός συστήματος κοινή έκδοσης ευρωπαϊκών αξιογράφων και ευρωομολόγων δυνάμει του άρθρου 85 του κανονισμού μέσα στα πλαίσια της ενίσχυσης της εποπτείας στην Ευρωζώνη. Αυτά τα ευρωπαϊκά αξιόγραφα θα ενισχύσουν την δημοσιονομική πειθαρχία και τις ευρωπαϊκές αγορές για να υπάρχει μεγαλύτερη ρευστότητα και τα κράτη-μέλη να έχουν μεγαλύτερη ε, πιστοληπτική, πιστοληπτικές δυνατότητες. Εάν υπάρχουν, ε, στη συνέχεια θα υπάρξει και μία πρόταση νομοθετικού περιεχομένου δυνάμει της ε, εφαρμογής αυτής της έκθεσης θα αναθεωρήσουμε και τους οποιοδήποτε μεθεπόμενους μηχανισμούς μέσα στα πλαίσια του Ταμείου Χρηματοοικονομικής Σταθερότητας. Αυτή η αναθεώρηση θα αποτιμήσει τον μηχανισμό χρηματοοικονομικής σταθερότητας για τη σταθερότητα της Ευρωζώνης και την ενίσχυση δημοσιονομικής πειθαρχίας μεταξύ κρατών μελών, καθώς και για την βελτίωση της χρηματοοικονομικής διακυβέρνησης και οικονομικής διακυβέρνησης. Επίσης θα ενισχύσουμε τις ε, μεταρρυθμίσεις που διέπουν το χρηματοπιστωτικό μηχανισμό για ενδεχόμενα ευεργετήματα και αποτελεσματικότητα, καθώς και τη λογοδοσία των διαφόρων θεσμικών οργάνων. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε τον... Ψηφίζουμε λοιπόν τώρα. Τροπολογία 10. Ψηφίσατε όλοι, έληξη ψηφοφορία αποτελέσματα εγκεκριμένα. Εγκρίθηκε. Ονομαστική ε, ψηφοφορία τώρα. Αρχίζουμε. Ψηφίσατε όλοι. Λήξη ψηφοφορίας. Εγκρίθηκε. Προχωράμε τώρα στο ψήφισμα νομοθετικού περιεχομένου. Τροπολογία 11. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίθηκε. Τροποποιημένη. Πρόταση. Υπέρ. Α, με συγχωρείτε. Ψηφίζουμε ονομαστικά. Ψηφίσατε όλοι. Λήξη ψηφοφορίας. Εγκρίθηκε. Σας ευχαριστώ και συγχαίρω την κυρία Γκουλάρα. Προχωράμε λοιπόν τώρα και θα ψηφίσουμε τα κατασταλτικά μέτρα για τη διόρθωση υπερβολικών μακροοικονομικών ανισορροπιών. Έκθεση Καρλ Χούγκλαντ, τροπολογία 4. Ψηφίζουμε. Ψηφίσατε. Λήξη της ψηφοφορίας. Εγκρίθηκε. Και τώρα ψηφίζουμε την τροποποιημένη πρότασία, πρόταση, με συγχωρείτε, ονομαστικά. Ψηφίσατε. Λήξη της ψηφοφορίας. Εγκρίθηκε. Εδώ έχουμε μία νομοθετική πρόταση, ονομαστική, ψηφοφορία παρακαλώ. Ψηφίσατε όλοι. Λήξη τη ψηφοφορία. Εγκρίθηκε. Ευχαριστώ πολύ και συγχαίρω βεβαίω τον κύριο Χάγκλαντ. Περνάμε λοιπόν τώρα στην έκθεση Ελίζα Φερέιρα πρόληψη και διόρθωση των υπερβολικών μακροοικονομικών ανισορροπιών. Η Κομισιόν ζήτησε το λόγο για να παρουσιάσει μία δήλωση. Ο Επίτροπος Ολυρέν έχει λοιπόν το λόγο. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε, αγαπητά μέλη, αξιότιμα μέλη. Θα ήθελα να κάνω την εξής δήλωση εκ μέρους της Κομισιόν. Η Κομισιόν καλωσορίζει την έγκριση του κανονισμού για την πρόληψη και τη διόρθωση των μακροοικονομικών ανισορροπιών. Ο κανονισμός αυτός αναγνωρίζει ότι τη φύση και του ενεπίγοντα χαρακτήρα και την πρόκληση και οι προκλήσεις μπορεί να διαφέρουν σημαντικά ανάλογα με το ε, ε, κράτος για το οποίο πρόκειται. Υπάρχει και ο βαθμός ε, του ευάλωτος και ο βαθμός προσαρμογής που απαιτείται και γι' αυτό είναι επίγον να ληφθούν μέτρα στα κράτη-μέλη τα οποία έχουν μεγάλα ελλείμματα στους τρέχοντες λογαριασμούς και έχουν και απώλεια ανταγωνιστικότητας. Επίσης, τα κράτη τα οποία ε, έχουν μεγάλα πλεονάσματα σε αυτόν τον τομέα θα πρέπει να λάβουν μέτρα ώστε να ενισχύσουν την εσωτερική ζήτηση και το δυναμικό ανάπτυξης. Κατά την εφαρμογή του κανονισμού, η Κομισιόν δεσμεύεται να σεβαστεί αυτές τις προσεγγίσεις και να εξασφαλίσει την εποπτεία τη μακροοικονομική ε, και για τα κράτη με ελλείμματα και για τα κράτη με πλεονάσματα κάνοντας τη σωστή διαφαροποίηση όσον αφορά τον επίγοντα χαρακτήρα και ε, των διορθωτικών μέτρων που πρέπει να ληφθούν. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, ευχαριστώ τον Επίτροπο και τώρα ψηφίζουμε τροπολογία 3, ονομοστική ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Λήξη ψηφοφορίας. Εγκρίθηκε. Και τώρα ψηφίζουμε την τροποποιημένη πρόταση, ονομαστική ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Έληξη ψηφοφορία. Εγκρίθηκε. Και προχωράμε τώρα στην ψηφοφορία του, της νομοθετικής πρότασης, τροπολογία 4. Υπέρ, σηκώστε το χέρι σας παρακαλώ, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίθηκε. Τώρα περνάμε στην ψηφοφορία της τροποποιημένης νομοθετικής πρότασης, ονομαστική ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι, λήξη ψηφοφορίας, Ευχαριστώ πολύ και συγχαίρω την κυρία Ελίσσα Φερέρα. Τώρα περνάμε στην έκθεση Διόγκο Φέιο σε σχέση με την εφαρμογή της διαδικασίας προβολικού ελλείμματος. Τροπολογία 7. Ψηφίζουμε. Ονομαστική ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Λήξη της ψηφοφορίας. Εγκρίθηκε. Και τώρα ψηφίζουμε την τροποποιημένη πρόταση. Ψηφίζουμε. Ψηφίσατε όλοι. Λήξη της ψηφοφορίας. Εγκρίθηκε. Και τώρα θα ψηφίσουμε για το νομοθετικό ψήφισμα. Ονομαστικά παρακαλώ. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Ευχαριστώ. Λήξη της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Συγχαίρω τον κύριο Φέιο. Και τώρα περνάμε στην έκθεση Vicky Ford, απαιτήσει για τα δημοσιονομικά πλαίσιο των κρατών μελών. Η Κομισιόν θέλει να κάνει μια δήλωση. Ο Επίτροπος Όλη δεν έχει το λόγο. Όπως εγκρίθηκε από την Κομισιόν είναι η δήλωση η Κομισιόν υπενθυμίζει την υποχρέωσή της και τη δέσμευσή της να εξασφαλίσει τα κράτη-μέλη να ε, συντάξουν ε, ε, πίνακες συσχετισμού με βάση την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα τις ανακοινώσουν ως προς τη μεταγραφή των νομοθετημάτων. Αυτά για να υπάρξει μεγαλύτερη νομοθετική διαφάνεια. Επίσης, θα εξετάσουμε και τη συμβατότητα εθνικών διατάξεων με κοινοτικέ. Λυπάμαι που δεν υπήρξε υποστήριξη για την πρόταση κανονισμού ε, για συγκεκριμένες απαιτήσει σε σχέση με τα δημοσιονομικά πλαίσια των κρατών μελών. Οι και συσχετισμού ε, θα έπρεπε να είναι υποχρεωτική. Συμβιβαστικά η Κομισιόν και για να εξασφαλίσει και την άμεση ε, υιοθέτηση αυτής της πρότασης δέχεται να αντικατασταθεί η υποχρέωση αυτών των, για, αυτούς τους πινά, πίνακες με μία διάταξη που παροτρύνει τα κράτη-μέλη να ε, χρησιμοποιήσουν αυτή την πρακτική. Η θέση της Κομισιόν όμως για αυτόν το φάκελο δεν θα θεωρηθεί σαν προηγούμενο Δηλαδή θα συνεχίσει η Κομισιόν τις προσπάθειες της για να βρει μαζί με το Συμβούλιο και το Ευρωκοινοβούλιο σωστή λύση σε αυτό το οριζόντιο θεσμικό ζήτημα. Ευχαριστώ τον Επίτροπο και τώρα περνάμε στην ψηφοφορία. Τροπολογία 3 με 5 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίθηκαν. Το σύνολο. Το τροποποιημένο σύνολο. Ψηφίζουμε. Ψηφίσατε όλοι. Έληξη ψηφοφορία. Εγκρίθηκε. Σας ευχαριστώ πολύ και συγχαίρω την κυρία Βίκη Φόρντ για το, την εργασία της. Κυρίες και κύριοι, έχουμε οριστικοποιήσει τις τροπολογίες, τις ψηφοφορίες για το Six Pack και θα ήθελα να συγχαρώ όλους τους ηγητές και την Επιτροπή Οικονομικών καθώς και όλες τις επιτροπές που υπέβαλαν γνωμοδοτήσεις σε σχέση με αυτές τις εκθέσεις. Πιστεύω ότι πραγματικά έγινε ένα μεγάλο έργο και θα ήθελα να τους ευχαριστήσω όλους θερμότατα. Το αποτέλεσμα είναι πολύ καλό και συγχαίρω όλα τα μέλη. Τώρα, συνεχίζει η ημερήσια διάταξη και περνάμε στον γενετήσιο προσανατολισμό και ταυτότητα του φίλου στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, παράγραφος 1. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίθηκε. Τροπολογία 12. Υπέρ, Kto jest przeciw? Νομίζω θα πρέπει να κάνουμε ένα ηλεκτρονικό έλεγχο. Παρακαλώ. Ψήφισαν όλοι πέρα στις ψηφοφορίες. Απορρίπτεται. Τροπολογία 1. Υπέρ. Κατά. Εποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 18. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 19. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Παράγραφος 8. Υπέρ. Κατά. Εποχές. Εγκρίνεται. Παράγραφος 9. Σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Εποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 20. Υπέρ. Κατά. Αποχές. απορρίπτωτο Να ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Τροπολογία 20. Ηλεκτρονικός έλεγχος. Czy wszyscy głosowali? Zamykam głosowanie. Ψήφισαν όλοι πέρα τη ψηφοφορία. Απορρίπτω. Τρει ταυτόσιμε τροπολογίε, 2, 7 και 14. Υπέρ. Κατά. Να ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Άρχη ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Πέρα τη ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Παρακαλώ σηκώντε τα χέρια σας ψηλά, αλλιώς δεν σας βλέπω. Τροπολογία 22, υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτω. 3, 9 και 16. Ταυτόσιμες υπέρ. Κατά. Να ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Η 3, 9 και 16 παρακαλώ. Ψήφισαν όλοι. Πέρα τη πληροφορία. Εγκρίνεται. Εγκρίνονται. Τροπολογίες 4, 8 και 15. Ταυτόσιμες. Υπέρ. Παρακαλώ ψηλά τα χέρια. Δεν σας βλέπω. Κατά. Να ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Ψήφισαν όλοι. Πέρας ψηφοφορίας. Ενεκρίθησαν. Τροπολογία 11 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 21 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται να ελέγξουμε αν θέλετε Έχει ψηφορία. τροπολογία 21 ψήφισαν όλοι Πέρας ψηφοφορίας. Ανακρίθηκε. Παράγραφος 12. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 5. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τρεις ταυτόσιμες τροπολογίες. Έξι, δέκα και δεκαεπτά. Υπέρ. Κατά. Επαθές Εγκρίνονται. Δεκατρία. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Λογική σκέψη Β. Στο προήμιο. Να ελέγξουμε. Θεώρηση 13 είχαμε. Άρχισε ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Πέρασε ψηφοφορία. Εγκρίνω. Ιδεολογική σκέψη Β. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 13 υπέρ. Κατά. Να ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Άρχη ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. πέρα ψηφοφορίας. Odrzucona. Ξεκάθαρα. Κοινό πρόταση νομοθετικού ψηφίσματος με ονομαστική κλίση η οποία έρχεται. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας ψηφοφορίας. Ενεκρίθη. Συγχαρητήρια.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 Περνάμε στι επεξηγήσει ψήφου. Επί της έκθεσης ε, Βόρτμαν Κόλ. Το λόγο έχει η κυρία Μανέσκου για ένα λεπτό. Ψήφισε υπέρ.